El señor Αγαπητές φίλες και φίλοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ξεκινήσουμε τις συνεδρίες. Το πρώτο σημείο είναι η έκθεση Γκέρινγκερ Ντεότεμπερ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Γκέριγκερ. Έχει έξι λεπτά η κυρία Γκέριγκερ Ντεότενμπεργκ στη διάθεσή της, τέσσερα λεπτά στην πρώτη φάση και δύο λεπτά εκ των υστέρων. Αυτό είναι μια σύσταση βέβαια, να μιλήσετε τέσσερα λεπτά στην πρωτολογία σας και μετά να ακολουθήσουν άλλα δύο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο πλαίσιο της ε, επικουρικότητας ε, θα πρέπει βέβαια να βελτιώσουμε την νομοθεσία, θα πρέπει η νομοθεσία να είναι